συναδέλφους τώρα να κάνουν τις επεξηγήσεις ψήφους, του, ψήφους των. Παρακαλώ. Καταρχήν όσον αφορά την έκθεση Φερνάντες, ε, ο συνάδελφος Πόσπισιλ παρακαλώ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 Ε, ελπίζω να πόρει μας ε, στην ε, Τσεχία έχουμε πολύ περισσότερα κονδύλια για τις πολιτικές ασφάλειας και μετανάστευσης και σε αυτό τη χρονική στιγμή χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων όπως και υπηρεσίες όπως τη Frontex χωρίς περισσότερα κονδύλια δεν θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μια ασφαλή Ευρώπη. Επίσης υπάρχει μια αύξηση κονδυλίων ε, για την εκπαίδευση των νέων που κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ε, πρόκειται για το πρόγραμμα Εράσμος. Η εκπαίδευση είναι από τους καλύτερους τρόπους να δείξουμε στη νέα γενεά ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι πολύ ευεργετική. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Πόσπιση. Δεν βλέπω τον συνάδελφο Πόρτσακ. Ο συνάδελφος Γιάρ τώρα. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν χαίρομαι ότι ε, επιβεβαιώθηκε ο προϋπολογισμός 2016 για να εργαστούμε όπως πρέπει. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας θέλω κάποια παράπονα να εκφράσω διότι όσον αφορά την Επιτροπή Προϋπολογισμών Όλε τι προτάσει τη Επιτροπής Γεωργίας τι απέρριψε. Όχι μόνο εκείνες που θα κόστιζαν κάποια κονδύλια, αλλά και εκείνες τις τροπολογίες και προτάσει που δεν θα συνεπαγόντουσαν πληρωμή κονδυλίων. Και αυτό με ενόχλησε. Θέλω οι συνάδελφοι λίγο πιο σοβαρά τι καλέ προτάσει τη Επιτροπής Γεωργίας να τι εξετάζουν και να τι αξιολογούν και να τι εγκρίνουν. Και έτσι η έγκριση του προπολογισμού θα είναι κάτι ευκολότερο μελλοντικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφε. Ο συνάδελφο Μάνικιν παρακαλώ. Μάνικινς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μέσω της ψήφισης ε, και έγκρισης ε, του προϋπολογισμού 2016 αυτό που συμβαίνει είναι το ότι εμείς ε, έχουμε και πιο αποτελεσματική χρήση κονδυλίων που εγκρίναμε μέσω των διαδικασιών. Αυτό υπερψηφίσαμε. Και το άρθρο 36 τι προβλέπει προβλέπει ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, τουλάχιστον τρεις φορές ε, θα πρέπει να διαβουλεύονται για την πιο αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Αυτό μπορούμε να το χαιρετήσουμε ως διαδικασία, ως πρόταση θα έχουμε μια πιο σε τακτά διαστήματα αναθεώρηση του τι συμβαίνει με τον προϋπολογισμό για να δούμε κατά πόσον οι στόχοι μπορούν να επιτεθούν και συνάδουν τα μέσα για την επιτεύξη των στόχων. Το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Κοινωνικό Ταμείο δυστυχώς πρέπει να πω <clears throat> υπέστησαν περικοπές στα κονδύλια τους. Αυτό δεν είναι θετικό. Όμως συνολικά υπάρχουν θετικές πτυχές στον προϋπολογισμό, γι' αυτό υπερψήφισα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. συνέχεια και ο συνάδελφος ε, Χάναν. Αποσύρει την παρέμβασή του. Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσει ψήφου για αυτήν την έκθεση. Περνάμε στι επεξηγήσει ψήφου στην έκθεση Φερέρα. Ο συνάδελφο Κόλτσακ, παρακαλώ. Δεν τον βλέπω στην αίθουσα, δεν ναι, παρίσταται. Ο συνάδελφο Γιάρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα να επενέσω όπως πρέπει την Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για εξαιρετική έκθεση πολλοί συμφωνούσαν, ούτως ή άλλως συμφώνησαν για το ότι η έκθεση αυτή υπερβολικά λέει έχει πολιτικό βάρος, πολιτικές τάσεις. Όμως είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα και όταν έχουμε θέματα φορολογίας και φορολογικής ε, δικαιοσύνης τα θέματα πρέπει να τύχουν παρακολούθησης από πλευράς μας. Προσβλέπω λοιπόν σε αυτό το έργο ε, σε σχέση με την κοινοβουλευτική μας επιτροπή και σε θετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Γιάρο. Συνάδελφος Κέλλη παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι έγινε ήδη πολύ καλή εργασία δουλειά από την Προεδρία ε, Σπίτι Γκονζάλες ίσω ο Αντιπρόεδρος αλλά βεβαίω ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό. Σε σχέση με αυτήν την ψηφοφορία λυπούμε ε, και είναι ασύνηθε για μας η Φίνεγκαν PPP. Εμείς ψηφίσαμε κατά ε, των μέτρων ε, και κατά της έκθεσης που είναι ασύνηθες διότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και πιστεύουμε ότι ξεπερνάει τα όρια ε, και ζητά από την από την Επιτροπή να κάνει ορισμένες έρευνες τώρα. Επίσης, η φορολογία είναι εθνικής αρμοδιότητας και αυτό έχει αναγνωριστεί παντού και πιστεύουμε ότι είναι ε, δεν είναι να περάσουμε στο CCCTB, δεν είναι προς το συμφέρον μας και γι' αυτό ψηφίσαμε κατά υπάρχουν πολύ καλά μέτρα μέσα σε αυτή. Νομίζω ότι η έκθεση πάει προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. Ευχαριστούμε συνάδελφε Κέλλη. Στη συνέχεια ο κύριος Μαμικίνς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορώ να προσθέσω τη φωνή μου στη φωνή των συναδέλφων που το έργο σας ως προεδρεύοντα σε αυτή την Ολομέλεια το επένεσαν. Τώρα επί της ουσίας όμως για τα φορολογικά θέματα. Μια πραγματικά <clears throat> δίκαιη φορολογική πολιτική είναι ακρογωνιαίο θεμέλιο, ακρογωνιαίο θεμέλιο της ε, ε, οικονομικής σταθερότητας και υγείας μιας χώρας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι έχουμε. Δεν έχουμε τόσους, τόσο πλούσιους φυσικούς πόρους ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας χωρίς φόρους και χωρίς φορολόγηση. Ο φυσικός μας πλούτος δεν το επιτρέπει, δεν είναι τόσο πλούσιος. Έχουμε τον φόρο κύκλου εργασιών, διάφορους φόρους, χρειαζόμαστε αυτή τη φορολόγηση. Καθένας όμως ο οποίος εργάζεται θα πρέπει και εκείνος να ε, αμείβεται για το έργο του, για την εργασία του και να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα διαβίωσής του και τα έξοδα και τις ανάγκες της οικογένειας του και πρέπει να υποστηρίζεται μέσω του μισθού του και έτσι οι φόροι πρέπει να είναι προσιτοί, να είναι χαμηλοί για τους εργαζόμενους ιδιαίτερα δηλαδή. Συνολικά πρέπει να χαιρετήσουμε αυτό το έγγραφο γι' αυτό υπερψήφισα. Ευχαριστώ πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφε Μάμικης. Η συνάδελφος Μπόλαν δεν παρίσταται. Ο συνάδελφος Πόσπισιλ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αποφάσισα να μην υποστηρίξω την έκθεση και έκανα αποχή. Τους λόγους τους εξήγησε ο προλαλής σας. Είναι πολύ δύσκολο να προωθήσουμε το CCTB ε, σε άμεσους φόρους, ειδικά στους εταιρικούς ε, φόρους. Εγώ ψηφίζω ένα κεντροδεξιό, ανήκω σε ένα κεντροδεξιό κόμμα και στο μανιφέστο του είναι να μην ενοποιηθεί η φορολογική βάση στην άμεση φορολογία και πρέπει να τηρήσω τις υποσχέσεις μου. Το να υποστηρίξω την αυτονομία στην άμεση φορολογία ε, των 100 μελών είναι πολύ σημαντικό. Ο υγιής ανταγωνισμός των διαφόρων φορολογικών ε, συστημάτων των 100 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω ότι είναι αποφελής. Φυσικά θα πρέπει να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό ε, τύπου Λουξεμβούργου ας πούμε. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Πρόσπιση. Ο συνάδελφος Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Το βασικό εμπόδιο μια κυβέρνηση που θέλει να συγκεντρώσει φόρου είναι ο διεθνή ανταγωνισμό. Μπορείτε να αυξήσετε του φόρου μέχρι ενό σημείου, και τότε αρχίζουν ε, τα λεφτά να φεύγουν προς πιο φιλικές ε, χώρες με φιλικότερα ε, φορολογικά καθεστώτα. Και η μοντέρνα τεχνολογία διευκολύνει την κίνηση των κεφαλαίων παγκόσμια. Μπορούμε να παραπονεθούμε, μπορούμε να νομοθετήσουμε κατά, αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε εντελώ. Δεν μπορούμε να το παρεμποδίσουμε. Ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την απώλεια εσόδων ω αποτέλεσμα τη φοροαποφυγή είναι καθιστώντα το δικό μα φορολογικό καθεστώ πιο ελκυστικό. Και εδώ μπαίνω στο βασικό επιχείρημα κατά της φορολογικής εναρμόνισης. Όσο το κάνεις πιο ομοιόμορφο, πιο συγκεντρωτικό, τότε επιτρέπει στις ε, κυβερνήσεις να βοηθηθούν χωρίς να υπάρχουν ε, προβλήματα και έλεγχοι. Ε, όταν αρμονίσουμε τους φόρους, στην πραγματικότητα θα υπάρξει μια ε, κατάσταση προς τα κάτω, συμπίεση προς τα κάτω. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια και ολοκληρώνει ο συνάδελφος Άρνοτ. Ευχαριστώ. Αυτό μου δείχνει ότι υπάρχουν δύο τίμιες θέσεις εδώ σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα είσαι ομοσπονδιακού τύπου ας πούμε, κράτος ε, και θα συμφωνείς με την αρμόνιση φορολογίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τότε θέλεις μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό, μεγαλύτερες εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια τίμια θέση. Ε, βέβαια, εγώ δεν την συμμερίζομαι. Η άλλη τι μία θέση είναι να πεις ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο το Ηνωμένο Βασίλειο ως ανεξάρτητο κράτος ε, και ως η ε, πέμπτη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Θέλουμε εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θέλουμε ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Τι μια θέση και αυτή. Ο τρίτος δρόμος όμως είναι το να είσαι, α πούμε, ε, και στην Ευρώπη και αλλά να λειτουργεί ω τροχοπέδι. Δεν είναι τίμιο για το ε, Ηνωμένο Βασίλειο αυτό και σωστό απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ούτε και απέναντι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει να αποφασίσουμε. Είμαστε μέσα ή έξω τελικά. Πρόεδρο, Σα ευχαριστώ, συνάδελφε Άρνετ. Ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσει ψήφου στην έκθεση Φεραίρα και Τόερε. Πάμε τώρα στην έκθεση επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση τη συναδέλφου Ντάτη που αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης Ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις. Γκονθάλεθ Πένια, παρακαλώ. Καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση διότι επικεντρώνεται στα συμπτώματα και όχι στα προβλήματα και στα αίτια του προβλήματος. Όλο το βάρος της έκθεσης αφορά περιοριστικά και καταστατικά μέτρα και τον κοινωνικό έλεγχο. Το πρόβλημα όμως του εξτρεμισμού, της ε, ε, επιδίνωσης των ελευθεριών μας ε, λαμβάνεται υπόψη. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα του φόβου δημιουργώντας περισσότερο φόβο και για τα κατεπήγοντα μέτρα έκτακτης κατάστασης για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και που ε, είχαμε το θέμα του Μάρτιν Σούλτς και της ε, Φεντερίκα Μογκερίνη τα αστυνομικά μέτρα ή καταστατικά μέτρα δεν επαρκούν μόνα τους για να ξεριζώσουμε, να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση πρέπει η κοινωνική ολοκλήρωση και ένταξη να προαχθεί ιδιαίτερα η εκπαίδευση και η μόρφωση ώστε να υπάρξουν εναλλακτικέ λύσεις για το μέλλον για μια κοινωνία που θα είναι συνεκτική και θα εκφράσει την αλληλεγγύη της. Θα είναι αλληλέγγυα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ συνάδελφε Γκονθάλεθ Πένια. Συνάδελφε Γκίλ, δεν σας βλέπω. Α, εδώ είσαστε συνάδελφε Γκίλ. Εντάξει, έχετε τον λόγο. Μπορείτε να παρέμβετε από όποιο μικρόφωνο επιθυμείτε. Thank Chair, and sorry. Ναι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Υποστήριξα την έκθεση αυτή επειδή πιστεύω ακράδοντα ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε ε, τις τρομοκρατικές οργανώσεις στο Ιράκ και στη Συρία δεν μπορούμε να αγνοούμε τα γεγονότα και να μην τα αντιμετωπίζουμε. Είτε πρόκειται για παστικοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο, στη Γαλλία ή στο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η πρόληψη και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για την ε, καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και ε, βεβαίως το θέμα αυτό δεν σταματάει στα εθνικά ε, σύνορα. Σκεφτείτε τα κοινωνικά δίκτυα, οι πλατφόρμες για άτομα που χειραγωγούν τους άλλους, που βρίσκονται απομονωμένοι από την υπόλοιπη κοινότητα. Είναι ένα θέμα που δεν αντιμετώπισαν τα κράτη-μέλη από μόνα τους. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το πράξει, να βρούμε λύση ε, χωρίς ε, να φύγουμε τις ελευθερίες ε, και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε στην κύριε. Ο συνάδελφος Μαύρου δεν Ο συνάδελφος Όμπερμαϊερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε οι τρομοκρατικές πράξεις στο Παρίσι ήταν, είναι οι πιο θλιβερές, κτρές πράξεις του Ισλαμικού εξ, ε, και δεν πρέπει κανείς να είναι ειδικό ε, για να προβλέψει να δει τις, ε, ε, Στην έκθεση αυτή όμως δεν αναφέρεται ούτε για στεναρότητα ούτε εντιμότητα τίποτα ντρεπόντουσαν φαίνεται να κατονομάσουν τα πράγματα, τον Ισλαμισμό δηλαδή στην Ευρώπη. Ε, όχι από εξτρεμιστές χριστιανούς ή Ιουδαίους, ε, Εβραίους ε, απειλούνται οι πολίτες της Ευρώπης σήμερα, αλλά από τους Ισλαμιστές. Αλλά δεν λέγεται αυτό, γιατί αυτό δεν είναι πολιτικά ορθό από ό,τι φαίνεται. Και δεν είχε το θάρρος η συγγήτρια να το πει αυτό. Για την ένωση, για τον ορισμό του εχθρού. Αν δεν υπάρχει στεναρότητα, τότε όταν μιλάμε για επανένταξη και τα λοιπά, χάσαμε ήδη τον πόλεμο και σηκώσαμε σηκώσαμε ψηλά τα χέρια και παραδοθήκαμε. σε ευχαριστώ συνάδελφε Ομπερμαϊα για την αποσαφήνιση σε σχέση με τον εισηγητή. Όπως είπατε πρόκειται για εισηγήτρια, εντάξει, το διορθώνω. Ακολουθεί ο συνάδελφος Πόσπιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, με χαρά υποστήριξα την εισήγηση αυτή, διότι πιστεύω ότι το πρόβλημα των ριζοσπαστικοποιημένων πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κράτη από μόνα τους δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν με 5.000 ζυχαντιστές μαχητές που θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν πηγή δυνητική τρομοκρατίας και κίνδυνο. Γι' αυτό χαίρομαι που έχουμε συγκεκριμένα ε, μέτρα στην έκθεση, δηλαδή οδηγία ε, σχετικά με κάτι που έχουμε εδώ και πολύ καιρό και που πρέπει να συμπληρωθεί και ελπίζω ότι θα είναι τομέας εγκληματικότητας εάν υπάρχει εκπαίδευση και ασκήσεις από τρομοκρατικές οργανώσεις και επίσης τα εξωτερικά σύνορα θα προστατευτούν καλύτερα. Γι' αυτό υποστήριξα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ συνάφη Πόσπισιφ. Τον συνάδελφο Πότσακ δεν τον βλέπω να παρίσταται. Ο συνάδελφος Σόγκορο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Το πρώτο ε, σημαντικό και σαφέσα από το Παρίσι είναι ε, το σύστημα ασφαλείας ε, και η κατάστατή του, ε, αν χρειαζόμαστε καλύτερα σύνορα, καλύτερα συστήματα πληροφοριών, προσβάσει στα δεδομένα των τρομοκρατών για να προστατεύσουμε τις ζωές των πολιτών. Είναι εξίσου σημαντικό για μας να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι αυτές οι σφαγές έγιναν από Ευρωπαίους πολίτες. Αν θέλουμε ο κόσμος να γίνει ασφαλέστερος θα πρέπει να αρχίσουμε με την κατανόηση του τι είναι αυτοί οι πολίτες που γίνονται εξτρεμιστές και σκοτώνουν ζωές στη χώρα τους και αλλού. Είναι εξτρεμιστές όπως λέχθηκε από τον επικεφαλής μιας, ενός ε, Ινστιτούτου στο Βέλγιο, στο Βίλ Βόρντε για την καταπολέμηση. Αν θέλουμε να αποτρέψουμε περισσότερα άτομα από το να πέσουν στα χέρια των τρομοκρατικών οργανώσεων, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς με την οικογένεια και την κοινωνία, διότι αυτούς τους δεσμούς προσπαθούν να διαρρήξουν οι στρατολογητές. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο συνάδελφος Γιάρ, παρακαλώ. Οι αριθμοί είναι φρικτοί και μας κάνουν και τρομάζουμε. 5.000 Ευρωπαίοι μάχονται στο Ιράκ και στη Συρία κατά των δικών μας αξιών και αρχών. Έχουν ε, ανατραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Θέλουν να αλλάξουν πράγματα δημοκρατικά που δεν τους αρέσουν, όμως επέλεξαν την τρομοκρατία για να το πράξουν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Η έκθεση είναι ισόρροπη και πρέπει φυσικά οι κοινωνικοί όροι και προϋποθέσεις να βελτιωθούν. Από την άλλη πλευρά όμως γνωρίζουμε, ακόμα και αν τα έχουν διευθετηθεί λυθεί τα κοινωνικά θέματα και έχουν ε, αποκατασταθεί η κακία ή το κακό ανήκει στον άνθρωπο ως χαρακτηριστικό και πρέπει να δούμε όλες τις δυνατότητες για να καταπολεμήσουμε την κακία και το έγκλημα. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση, χρειάζονται ευρωπαϊκές λύσεις. Γι' αυτό η παράκλησή μου. Εκθέσεις έχουμε, αρκετές έχουμε συντάξει. Παρακαλώ επιτέλους τα κράτη-μέλη να διαθέσουν τα αναγκαία κονδύλια ώστε να προχωρήσουμε στις πράξεις, στη δράση. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Ακολουθεί ο συνάδελφο Κέλλη. Ε, ε, Αυτή ψηφίσαμε με την ομάδα μα και βεβαίω υπέρ της ίδιας της έκθεσης. Χωρίς αναμφισβήτητα οι επιθέσεις στο Παρίσι μας έδειξαν ότι όλοι κινδυνεύουμε, όλοι μας στον κόσμο στον δυτικό κόσμο. Είμαστε στόχος ε, του ISIS και το είδαμε σε βίντεο ε, τα οποία δημοσιεύτηκαν. Μιλάνε για ε, για την, τους διαβόλους και αναφέρουν 60 χώρες μεταξύ των οποίων και η δική μου. Πρέπει λοιπόν να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να είμαστε ενωμένοι, να εργαστούμε σκληρά εναντίον της μάστιγας αυτής και κυρίως θα πρέπει να ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και με χαρά είδα ότι 630 ε, ψήφισαν υπέρ. Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Κέλλη. Ο συνάδελφος Νέκοφ ακολουθεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι τελευταίες επιθέσεις στο Παρίσι και στο Μαλί δείχνουν ότι η τρομοκρατία δεν έχει σύνορα. Θα πρέπει να δράσουμε παγκόσμια και ενωμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω τη σύμβαση του Παρισιού, τη σύνοδο του Παρισιού των Υπουργών όπου θα επικεντρώσουν στις ανθρώπινες αξίες όπως ελευθερία, καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης ε, από πολύ νεαρή ηλικία. Η Ευρώπη περνάει δύσκολες στιγμές. Θα πρέπει η εκπαίδευση να αφορά όλους, να μην αποκλείει κανένα, να δημιουργούνται μέσω αυτής ε, υπεύθυνοι πολίτε, ε, με ανεκτικότητα, ε, με κριτική σκέψη και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εστιάσουν σε αυτό, ούτω ώστε να μάθουν να κρίνουν την ποιότητα των πληροφοριών και στο ίντερνετ και να είναι λιγότερο ευάλωτοι σε τέτοια μηνύματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε συνάδελφε Νέκοφ. Ο συνάδελφο Μαμικίν, παρακαλώ ακολουθεί. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι πολύ απλό. Γιατί το Βέλγιο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν για τους τρομοκράτες την αιστεία ή τη βάση τους, την έδρα τους. Η Ευρώπη ουσιαστικά έχει τις δικές της αξίες και γίνεται θύμα των δικών της αρχών και αξιών. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι τρομοκράτες τις δικές μας αρχές και αξίες ε, να τις ε, εκμεταλλευτούν ώστε να ξεκινήσουν τέτοιου είδους τρομοκρατικά πλήγματα. Πρέπει τα σύνορά μας ε, να διασφαλιστούν διότι αν δεν υπάρχει ασφάλεια έχουμε τέτοιου είδους τρομοκρατικά πλήγματα σαν αυτά που βιώσαμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι οι μυστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία καλύτερα μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Μάμικιν. Σας συνάδελφος Χάναν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν θέλουμε οι έπικοι και τα παιδιά τους να ενταχθούν, οι άπικοι, θα πρέπει να τους προσφέρουμε κάτι. Θα πρέπει να τους να σημαίζονται και αυτοί τον πατριωτισμό, να έχουν κοινέ αξίες, ε, με τους πολίτες μας. Ε, αυτοί που μεγαλώνουν στην Ευρώπη βλέπουν ότι έχουμε τα κράτη-έθνη. Φανταστείτε ένα παιδί, ας πούμε μαροκινής ε, καταγωγής που μεγαλώνει στο Μόλεμπεκ. Ποια είναι η εμπειρία του. Ε, έρχεται σε επαφή με ένα κράτος ε, το οποίο του μάθανε να το μισεί. βλέπει τις δύο γλωσσικές κοινότητες στο Βέλγιο, οι οποίες ε, η κάθε μία είναι στραμμένη προς το εσωτερικό της και δεν υπάρχει καμία ε, αλληλεπίδραση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. θα πρέπει η, η αίσθηση τη ταυτότητα να είναι πολύ πιο έντονη, α πούμε. Ε, για να αντιμετωπίσουμε την, ε, τον Ισλαμισμό θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε... Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε συνάδελφε Κόμπερν. Ε, Δεν επιτίθεμαι σε εσά, αλλά στο σύστημα, πρόεδρε, θέλω να πω καταρχά, ε, που κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και το τρομοκρατικό είναι ότι η νόμοι στην Ευρώπη και ελευθερίες ε, έρονται τόσο γρήγορα ε, που μου, μου έρχεται στο μυαλό ας πούμε η δημοπρασία και το πώς αλλάζουν οι τιμές ε, η μία μετά την άλλη. Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι και όχι ταχύτεροι. Οι αριστεροί και οι φιλελεύθεροι επίσης ε, καλύπτουν τα λάθη τους ανοίγοντας την πόρτα στην μετανάστευση. με αυταρχική ε, νομοθεσία κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουμε έτσι τους ε, εγκληματίες. Το τραγικό και η απειλή είναι η ταχύτητα με την οποία περνάνε νέοι νόμοι. Και δεύτερον, το πρόβλημα της αριστεράς, η οποία προσπαθεί να καλύψει τα λάθη της με αυταρχικούς νόμους. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο συνάδελφος Άρνοτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πράξη αυτές έχουμε στα σχολεία μια ουδέτερη πρόπτικη και έχω μια ανησυχία για αυτήν την έκθεση. Είχαμε μια τροπολογία μετά την παράγραφο 25 νομίντο λέγοντας ότι η καθήκοντα των ε, κρατών μελών είναι να εξασφαλίσουν εκπαιδευτικά ε, συστήματα προώθησης αξιών και αρχών. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ευθύνη ε, της, του, του Βρετανικού κράτους να πολιτικοποιεί έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα. Ε, θα πρέπει να εκπαιδεύονται τα παιδιά σε δεξιότητες για να έχουν προσόντα και όχι για το τι πρέπει να σκέφτονται. Βεβαίως, ε, οι αξίες αυτές ε, δεν ξέρω τι είναι και γι' αυτό αισθάνθηκα ότι έπρεπε να ψηφίσω εναντίον της έκθεσης αυτής. Σας ευχαριστούμε για να ολοκληρώσει τις επεξηγήσεις ψήφου αυτή την έκθεση ο κύριος Έθριτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ψήφισα κατά μια έκθεση για την πρόληψη της ρίζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατίας στην Ευρώπη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ικανή να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, μας λέει. Είχαμε ένα σωρό συζητήσεις είτε είμαστε φτωχοί, είτε δεν έχουμε την ευκαιρία, είτε είμαστε ε, σκληροί διότι μιλάμε κατά της μετανάστευσης. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τους λόγους και πάντοτε χάνουμε την ουσία, επειδή ε, ε, διάφοροι θα το δουν αυτό και δείχνουμε το δρόμο και ε, βλέπουμε ότι η μαζική μετανάστευση έχει να κάνει κάτι με αυτό το φαινόμενο. Μεταφέρουμε ε, χιλιάδες άτομα που δεν ξέρουμε τι σχέση έχουν. Και σε αυτή τη συζήτηση είχαμε μια ψηφοφορία όπου πολλοί δεν ξέρανε γιατί ψήφιζαν. Νομίζω ότι δεν έχει καμία ουσία, κανένα νόημα αυτή η έκθεση. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε συνάδελφε Ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Ντάτι. Ακολουθούν οι επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Κρίστενσεν για το στρατηγικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την περίοδο 2014-2020. <clears throat> Η συνάδελφος Γκονθάλετ Πένια έχει τον λόγο παρακαλώ συμφωνούμε με τη διάγνωση που κάνει αυτή η έκθεση, την αστάθεια στην απασχόληση, χαμηλούς μισθούς, αδιάκριτη, ε, χωρίς όρους ε, πρόσληψη, επισφαλής εργασία. Είναι συντελεστές που συνεισφέρουν στην επιδείνωση της υγείας ε, και των εργαζομένων και των γυναικών και ανδρών. Όταν δεν είναι δεν είναι εντάξει μια επιχείρηση στα καθήκοντά της έχουμε δράματα όπως ε, τον δηλητηριασμό από υδράργυρο όπως ε, στην Αστούρια ε, συνέβη σε μια επιχείρηση στο τέλος τα σπασμένα τα πληρώνουμε όλοι μας με απώλεια παραγωγικότητας των οικονομιών μας και μεγαλύτερες δαπάνες για τα εθνικά συστήματα υγείας μας και κοινωνικής περίθαλψης επίσης και για την εστίαση στα φύλλα, στο θέμα των φύλων στην Ευρώπη θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ξεχωρίσουμε καθορίσουμε τα πράγματα αντί να επιβαρύνονται οι γυναίκες με διπλή και τριπλή υποχρέωση και εργασία. Και έχουμε θετικά στοιχεία όμως επίσης θέλουμε να απευθύνουμε μια προειδοποίηση στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές διότι συνέχισαν να, να υποστηρίζουν τις πολιτικές λιτότητας και αυτό σημαίνει ότι διακόπτεται από το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο συνάδελφος Σούλτσε. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό και σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλειοψηφία των 217 εκατομμυρίων εργαζομένων γυναικών και ανδρών να δημιουργήσει ένα νέο καλύτερο πλαίσιο για την υγεία τους και την ασφάλειά τους από το 2014 στο 2020. Για μένα ήταν αποφασιστική σημασία σε αυτό. Η πρόληψη όσον αφορά ε, ασθένειες που προκαλούνται από την εργασία και η εφαρμογή των κανονισμών και κανόνων με καλύτερο τρόπο είναι σημαντικό η νομοθεσία για τα εργασιακά θέματα και την προστασία τη ε, εργασία και τη υγεία των εργαζομένων να μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα. Όταν τα επιτύχουμε όλα αυτά, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για καινούριου κανόνε και κανονισμού. Είναι οι επιχειρήσει οι οποίε πρέπει να προχωρήσουν, είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που πρέπει να προσαρμοστούν. Εγώ πιστεύω ότι οι βέλτιστε πρακτικέ και τα παραδείγματα που δίνονται στην έκθεση για την εφαρμογή στην οδηγία, εντάξει, συνολικά πιστεύω ότι μια σωστή ισορροπία έχει εξευρεθεί σε αυτή την έκθεση για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Γι' αυτό υπερψήφισα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε, συνάδελφε Σούλτσε. Ακολουθεί η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η επισφαλής διαμόρφωση εργασιακών μορφών, η άτακτη ρυθμή εργασίας, το επίπεδο ανακύκλωσης των συμβάσεων είναι συντελεστές που οδηγούν σε ατυχήματα και σε τέτοιες περιπτώσεις και ασθένειες. Στην Ισπανία εμείς έχουμε καταβάλει προσπάθειες. Ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα των συνδικάτων και για την εκπόνηση στρατηγικών για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Δεν είμαστε υπέρ να μειωθούν τα θέματα για τα εργασιακά από πλευρά των οργανώσεων. Μετά από αυτά θέλω να αναφερθώ στα ενδοκρινολογικά θέματα. Όσον αφορά την βούληση της ε, ρύθμισης της ε, υγείας ε, για τα θέματα που έχουν επιπτώσεις ενδοκρινολογικά μπορούν να οδηγήσουν σε κρίσεις οι καταστάσεις αυτές ενώ υπάρχουν αυτά τα, αυτές οι ουσίες σε κτίρια στην Ευρώπη. Ζητούμε να υπάρχει ένα πλαίσιο για την αποζημίωση των ε, εργαζομένων όσον αφορά την ασθένεια σιλικόσης για παράδειγμα. Τίποτα δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστούμε λέγει ο Πρόεδρος κυρία Λόπεθ Μπερμέχο, στη συνέχεια ο συνάδελφος Σόγκορ να αυξήσουμε την ασφάλεια στην υγεία δεν είναι προ το συμφέρον των εργαζομένων, αλλά προ το συμφέρον και των επιχειρήσεων και των οικονομιών, γιατί θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα κτλ. Και τα συστήματα περίθαλψης και πιστεύουμε ότι οι αποτελεσματικοί κανόνες ε, για την υγεία στον χώρο εργασία και αυστηρή εφαρμογή ανεξάρτητα από το μέγεθο τη επιχείρηση είναι σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη ειδικέ καταστάσει και ανάγκη, ε, τι ανάγκε ειδικών επιχειρήσεων και την παροχή ε, βοήθεια ε, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν την νομοθεσία για την ασφάλεια στην εργασία. Συμφωνώ με την έκκληση επίση ότι θα πρέπει να ε, αυξήσουμε τα μέτρα κατά τη αδήλωτη εργασία, γιατί οι αδήλωτοι εργαζόμενοι είναι οι πιο εκτεθειμένοι σε ατυχήματα στον χώρο εργασία. Ευχαριστώ. Προέδρο. σας ευχαριστούμε συνάδελφε Σόγκορ. Ακολουθεί ο συνάδελφο Γιάρ. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο συνάδελφο Σούτ στην επεξήγηση ψήφου μίλησε από την καρδιά μου και εξέφρασε τι απόψει μου. Είναι μια τυπική έκθεση που μπορεί κανείς να υπερψηφίσει. Όλα τα πράγματα που αναφέρονται είναι ορθά. Θέλουμε προστασία στην εργασία, στον χώρο εργασίας και προστασία της υγείας πανευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά και να είμαστε αποτελεσματικοί. Σωστό αυτό. Αλλά να μην οδηγηθούμε σε μια χιονοστιβάδα γραφειοκρατικών μέτρων που θα ισοπεδώσουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όταν μιλάμε για βέλτιστες πρακτικές δεν είναι οι βέλτισε πρακτικέ ε, στο προσώφερο τη γραφειοκρατία, αλλά για να είμαστε αποτελεσματικοί στο τέλο τέλο. και αυτό είναι μια προειδοποίηση που θέλω να δώσω στου αρμόδιου συναδέφου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να μεριμνήσουν το καλό που θέλουμε να πετύχουμε να μην υπονομευθεί με γραφειοκρατική χιονοστιβάδα που δεν θα, έχει, δεν θα δώσει κανένα αποτέλεσμα και θα αυξηθούν οι επιφυλάξει ε, για τέτοιου είδου ε, στόχου. Ευχαριστώ. ευχαριστώ Ευχαριστώ συνάδελφε Γιά. Ο συνάδελφος συναφεγιά. αυτό το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στη Σουηδία τα συνδικάτα μας και άλλοι φορείς έχουν λάβει σημαντική, σημαντικά μέτρα και έχουν συμμετέχει στις εθνικές αποφάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στην, εργασία. Το σουηδικό μοντέλο δεν θέλω να αποδυναμωθεί χώνοντα ε, τη μύτη της Ευρωπαϊκή Ένωση στις υποθέσεις μας. γι' αυτό καταψήφισα αυτή την πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θέλει να μπερδεύεται σε όλα ε, τα εθνικά θέματα. Ε, και δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο σπάνια υπάρχει βελτίωση. Αντίθετα μας φοράει ένα μοντέλο το ίδιο για όλους και οδηγεί αυτό στην καταστροφή. Εμείς είμαστε ηγέτες, ε, έχουμε ηγετικό ρόλο στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να το κρατήσουμε το μοντέλο μας και πιστεύουμε ότι αν δεχοθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα, κάνουμε, θα τα καταφέρουμε καλύτερα εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε. Λόγκρεν, ακολουθεί ο συνάδελφος Μαμικίνς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Γεωστρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας για το 2014-2020. Το στρατηγικό αυτό πλαίσιο είναι ένα έγγραφο το οποίο κατεπηγόντως χρειαζόμαστε. Κάνουμε λόγο για τους στόχους που μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας πρέπει να έχουν επιτευχθεί συνολικά. Νομικές πτυχές, ψυχολογικά ζητήματα, θέματα ανταγωνισμού, όλα πρέπει συνολικά να εξεταστούν για να προχωρήσουμε. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών μπορέσαμε και να μειώσουμε την ανεργία, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μια και έχουν όλοι οι άνθρωποι το δικαίωμα να εργάζονται στην εργασία και για να εργάζονται χρειάζονται και θετικούς καλούς όρους απασχόλησης στην εργασία τους. Στην Λετωνία, στη χώρα μου, πρέπει να πω ότι αυτό που βλέπουμε είναι θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τους αρνητικούς όρους απασχόληση και αυτό πρέπει, απασχόλησης και αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Ευχαριστούμε. Τον συνάδελφο Χάναν δεν τον βλέπω να παρίσταται, οπότε ολοκληρώθηκαν και οι υπεξηγήσεις ψήφου σε αυτή την έκθεση Κρίστενσεν. Και διακόπτουμε τη συνεδρίασή μας μέχρι τις 3, 15.00. Καλή όρεξη σε όλους σας. Στις 3 θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.